Okay, colleagues, um, we have reached uh, point Φτάσαμε στο σημείο 4. Κάναμε μια διακοπή για να περιμένουμε να έρθει ο συγητή. Χαίρομαι διότι κατέφθασε ο κ. Σόγκορ. Ευχαριστώ του συναδέλφου για την παρουσία του, Την πιστή του παρουσία. Εργάζονται σκληρά. Αναβλήθη η ψηφοφορία του πνευματικά δικαιώματα. Εκτιμώ το ότι είσαστε παρόντε για τα άλλα σημεία τη ημερήσια διατάξεω. Δεν θα μπορούσαμε να συζητήσουμε εν τη απουσία σα. Ευχαριστώ για την παρουσία σα. Πάμε. Σημείο 4. Έκθεση του 2017 για την Ευρωπαϊκή Ιθυγένεια να, να ισχυροποιήσουμε τα δικαιώματα των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. και ο κ. Σόγκορ. παρουσίασε του σχέδιου γνωμοδοτήσεως στην Επιτροπή Αναφορών 4 Σεπτεμβρίου. 118 τροπολογίες υπευλήθησαν όσον αφορά τη γνωμοδότηση και τώρα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε τι εν λόγω τροπολογίε υπενθύμηση. Ε, σύμφωνα με το άρθρο 54 συμμετέχουμε και εμείς στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Εξετάζουμε το θέμα απειλών κατά της ασφαλείας, προστασία των δικαιωμάτων των, ε, που έχουν ευρωπαϊκή ηθαγένεια και να στηρίξουμε και τα θύματα εγκληματικών ενεργειών. Ε, ο κύριος Σόγκο λοιπόν έχει το λόγο να μας κάνει μια παρουσίαση και Και ευχαριστώ Πρόεδρε, όπως ανέφερα στην παρουσίαση του σχεδίου εκθέσεως, η έννοια της ηθαγενείας ε, ε, δεν καλύτερο το πλήρως από την ε, γνωμοδότηση. Γι' αυτό τονώσαμε περισσότερο το κείμενο και εκφράζουμε λεπτομερέστερα την άποψή μας για το θέμα. 118 τροπολογίες έχουν υποβληθεί, αναφέρονται στην ασφάλεια, την προστασία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενώσης στο εξωτερικό και η προστασία των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών. Επίσης αναφέρονται και νέοι τομείς, μη διάκριση, ισότητα όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ένα παράδειγμα, ανεξάρτητα αν ανήκουν σε κάποια μειονοτική ομάδα. Οι περισσότερες τροπολογίες ακολουθούσαν αυτή την κατεύθυνση, κυρίως γινόταν αναφορά στην κατάσταση των αυτοχθόνων εθνοτικών μειονοτήτων, την ανησυχητική κατάσταση των Ρωμά, των ΛΟΑΔ, των ανθρώπων με αναπηρία και των ηλικιωμένων. Υπάρχει γενική συμφωνία μεταξύ μας. Τέτοιες ομάδες χρήζουν μεγαλύτερας προστασίας για να μην υπάρχει διάκριση και να υπάρχει ισότητα σύμφωνα με τις συνθήκες. Συμφωνούμε και επί άλλου ότι η θαγένεια δημιουργεί δικαιώματα. Πρέπει να επικρατεί το κάτω δικαίωμα δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και να υπάρχει ένα ισχυρό πλαίσιο που τα προστατεύει αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο τομέα. Brexit και τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Πολύ σημαντικό για εκατομμύρια πολιτών και τις δύο πλευρές της μάχης που αισθάνονται ε, ανασφάλεια και ανησυχία τώρα. Πολλοί τομεί καλύπτονται που δεν του ανέφερα. Ευχαριστώ του Κιώδη για την υποστήριξή του για τι διάφορε τροπολογίε και προσβλέπω σε μια αγαστή συνεργασία για τι συμβαστικέ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριο Σογκάρ. Κάποιος από τους σκιώδεις θέλει να μιλήσει. Ο κ. Βάντερ Χόζε. Θα ήθελα μόνο να ευχαριστήσω τον εισηγητή κ. Βάινταν Χέλσερ. Ήταν πολύ καλή η συνεργασία μας. Uh, Συζητήσαμε όλο το θέμα, ε, βρήκαμε συμβιβαστικές ε, λύσεις και πραγματικά πιστεύω ότι μπορούμε να ε, προχωρήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Είναι σημαντική η συνεισφορά της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Αλμπιόλη είναι σκιώδης από την Ενωτική Αριστερά. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του και να θέσω μερικά ζητήματα που θεωρούμε σημαντικά. Η γνωμοδότηση αυτή εγγράφεται στις προσπάθειες να σφυριλατηθεί μια κοινή ηθαγένεια για όλους τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό δεν έχει μεγάλο νόημα εάν παραγνωρίσουμε ε, τις ανισότητες που διαπερνούν ε, τις κοινωνίας μας. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για ηθαγένεια χωρίς να αναφέρουμε τις πολιτικές λιτότητας, περικοπών, ιδιωτικοποίησης κοινοφελών υπηρεσιών, όλα αυτά. Άρα αυτή είναι η ανισότητα στην πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, παιδεία, υγεία, ενέργεια. Για μας αυτά είναι δικαιώματα που θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν κάναμε κάποιες τροπολογίες. Στη συνέχεια πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι απορρίπτουμε περίτρανα το γεγονός ότι πολιτικές ασφαλείας σε πολλές περιπτώσεις περικόπτουν και καταστέλουν δικαιώματα των πολιτών, ανδρών και γυναικών. Επίτε, πλέον κάναμε μια τροπολογία που ζητούμε να απεμπλακεί η οδηγία κατά των διακρίσεων. Διότι θεωρούμε επίσης ότι αυτού του είδους οι διακρίσεις, η ε, ξενοφοβική βία, η ομοφοβία κτλ ε, επιθέσεις κατά τον ΛΟΑΔ είναι θέματα που έχουν να κάνουν με δικαιώματα ηθαγένειας. Και κάτι ακόμα. Υπάρχει ένα σημαντικό τμήμα των ανθρώπων που ζουν στην κοινωνία μας που δεν έχουν καν πρόσβαση σε καμία ηθαγένεια και δεν έχουν δικαιώματα. Υπολογίζεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν 11 εκατομμύρια ε, άνθρωποι ε, που είναι είτε απάτριδες είτε μετανάστες ε, χωρίς χαρτιά, χωρίς να νομιμοποιούν την παρουσία τους και δεν έχουν δικαίωμα σε τίποτα. Ε, εμείς θεωρούμε ότι όποιος ζει στα κράτη-μέλη μας θα πρέπει να είναι Ευρωπαίος πολίτης. Άρα να έχει όλα αυτά τα συμπαραμαρτούντα δικαιώματα. Τίποτα άλλο δεν έχω να προσθέσω. Αυτά, αυτές είναι οι τροπολογίες μας. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σόγκαρ, θέλετε να συνοψίσετε μήπως. Όχι. Φτάσαμε στο τέλος η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ στις 6 Νοεμβρίου. Οπότε, πάμε σε άλλο. Διάλειμμα. Τηλεφωνούμε στην κυρία Μπεσορέλ να δούμε αν θα καταφτάσει το ταχύτερο δυνατόν, ούτω ώστε να συζητήσουμε το επόμενο σημείο τη ημερησία διατάξεω. Λίγη υπομονή παρακαλώ. Λυπούμε. Ξέρω, είναι πέμπτη πρωί και θέλουμε να κινηθούμε τάχιστα ενοχλούμε τους πάντες τώρα, τους καταπιέζουμε όλους. Και στον κύριο Βόσο ακόμα τηλεφωνούμε να κάνει και αυτός προθέρμανση. Αυτά συμβαίνουν όταν δεν υπάρχει ψηφοφορία. Είναι μετάβλητη όλη η κατάσταση. If Αν φτάσει ο κύριος Βος πριν την κυρία Μπεσερέλ θα αλλάξουμε σειρά.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 Okay, um, Ας προχωρήσουμε. Είναι πέμπτη πρωί. Και πρέπει να προχωρήσουμε. Παρίστε τη συγκήτρια. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Σημείο 5. Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση προτάσεως οδηγίας για τις αστικά στοιχεία των ποινικών πράξεων και κυρώσεων στον τομέα των παράνομων, διακίνησης παράνομων ναρκωτικών και ορισμούς της ενίας ναρκωτικών. Όταν είναι έτοιμη η συγκήτρια, θα ασχοληθεί με τη θέση του Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση που υιοθετήθηκε τον Απρίλιο του 2014. Μετά σε διαπραγματεύσουν το Συμβούλιο και συμφωνία εγκρίναμε τη θέση στις 8 Ιουνίου σαν Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και η πρώτη κοινή θέση 25 Σεπτεμβρίου υιοθέτησε στο Συμβούλιο και αντικατοπτεί στη θέση του Κοινοβουλίου μετά από έλεγχο των αρμοδίων νομικών υπηρεσιών και των διαθεσμικών οργάνων. Το Κοινοβούλιο αναμένει αναμένεται θετήσει τη θέση του στην πρώτη ανάγνωση όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού στην επόμενη Ολομέλεια και ταυτόχρονα με την έγκριση τη οδηγία. Λοιπόν, Τερέζα, είσαι έτοιμη? Ναι, είμαι, λέει η Τερέζα. Συγγνώμη που σε πιέζω, πιέζω όλου. όχι λέει η Τερέζα, προείδρευα τη αντιπροσωπεία του Μεξικού και ήταν στην άλλη άκρη του χτιρίου. Νόμιζα ότι ήμασταν στι 11, θα συζητούσαμε στις 11. Ναι, το ξέρω, λέει ο Πρόεδρο, Ξέρω ότι και εσύ και ο κύριος Βόση είστε συνεδριάσεις. Κάποιοι του σκιώδη απουσιάζουν. Επειδή επειδή είναι πέμπτη πρωί πρέπει να προχωρήσουμε. Λοιπόν, σε παρακαλώ κάνε την παρουσίαση αν έχεις την καλοσύνη. Κάνε ένα πρόβλημα. Θα με ακούσουν οι παριστάμενοι. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η εξέταση του σχεδίου έκθεση σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση για την οδηγία των νέων ψυχοτρόπων ουσιών ε, θα ήθελα να κάνω μια μικρή επισκόπηση της διαδρομής που κάναμε μέχρι σήμερα, γιατί θεωρώ το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Οι νέες ψυχότροπες ε, ουσίες συνιστούν μια μεγάλη απειλή για την ε, υγεία και την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών, ιδιαίτερα για τους νέους. Κάθε χρόνο πολλοί νέοι, οι περισσότεροι από αυτούς άνδρες, πεθαίνουν μετά από τη χρήση ψυχότροπων ουσιών και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία κατά των ε, ναρκωτικών ανείχνευσε 509 ε, νέες ουσίες ε, πέρσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η τάση βαίνει αυξούμενη με απίστευτο τρόπο η αύξηση της πώληση μέσω ίντερνετ αυτού του τύπου ε, ναρκωτικών και η ευκολία να παραχθούν ε, παράνομα σε εργαστήρια ε, καταστά χέρις για την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει στην παραγωγή νέων ψυχότροπων ουσιών. Η απόφαση πλαίσιο του 2014 ήταν αποτελεσματική όσον αφορά την ανείχνευση αυτών των ουσιών. Γι' αυτό η Επιτροπή κατάρτισε με ένα νέο κανονισμό και κατά συνέπεια μια νέα οδηγία για να υπερβεί τη νομική πρόκληση. Και αυτός ο κανονισμός, αυτό το κανονισμό είχα ως ε, συνεργάτη τον κύριο Βόνη, ο οποίος ε, το κατήρτισε πέντε χρόνια αργότερα τελικά καταλήξαμε σε μια συμφωνία. Δεν ήταν εύκολο, αλλά το καταφέραμε. Αυτά τα δύο εργαλεία, η οδηγία και ο κανονισμός, όπως είπα, είχαν μια, ένα, μια μακρά διαδρομή. Και Καμία από τις ε, τριμερείς συναντήσεις δεν κατέληξε σε επιτυχία. Χάρη στην Προεδρία της Μάλτας ε, κατορθώσαμε μία συμφωνία στην, ε, όσον αφορά την οδηγία. Θεωρώ είναι μία επιτυχία για το σώμα μας γιατί συμπεριλήφθησαν πολλά από τα αιτήματά μας και θα αναφερθώ σε τρία για τα οποία αναγωνίστηκαμε πάρα πολύ στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου που αρχικά ήταν ε, δύσκολος γιατί το Συμβούλιο ήταν αρνητικό πρώταν ε, ε, κατεξουδότηση ε, πράξης. Το Κοινοβούλιο κατήρτισε το κείμενο της Επιτροπής ούτως ώστε να τις εγκρίνει, η, να τις υιοθετήσει η Επιτροπή. Μετά από μακρά συζήτηση ε, κατορθώσαμε να πετύχουμε τις κατεξουδότηση πράξης. Το δεύτερο πρόβλημα και εμπόδιο ήταν η το τμήμα 2 που αφορά την πρόταση του Συμβουλίου να εγκριθούν κατεξοδότηση πράξεις που θα ανατεθούν στην Επιτροπή για μια συγκεκριμένη περίοδο και χωρίς ε, πιθανότητα αναβολής. Εμείς ε, ε, προτιμούσαμε να υπάρξει διοργανική συμφωνία, δηλαδή να εφαρμοστούν οι της πράξη για μια ταυτόσιμη περίοδο εφαρμογής δηλαδή να διαφρυνθεί εφόσον ε, δεν ε, ε, υπάρξει αντίθετη άποψη. Τέλος, το Συμβούλιο συμφώνησε. Και το τελευταίο σημείο είναι ότι κατορθώσαμε να πετύχουμε μια συμφωνία για την πρόταση του Κοινοβουλίου να καταργηθεί η παράγραφος 3 του άρθρου 1 της οδηγίας. Αυτή η παράγραφος λέει ότι αν η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν είναι αναγκαίο να εγκριθεί μια, να υιοθετεί μια ε, πράξη όσον αφορά τη συμπερίληψη μιας ψυχοτρόπου ουσίας στην, ε, στα ναρκωτικά ε, μπορεί να γίνει με, ε, χωρίς κατεξόδευση πράξη και μετά από διαβουλεύσεις ε, με την Προεδρία της Μάλτας συμφώνησαν να διαγραφεί αυτή η παράγραφος η οποία ήταν πολύ σημαντική για το Κοινοβούλιο. Χάρη στην Προεδρία της Μάλτας ε, μπορέσαμε να πετύχουμε μια ισορροπία. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για το ρόλο που διαδραμάτισε σε αυτή την ε, συνάντηση και ιδιαίτερα στον κύριο Πόνη που συνέβαλε στην επίτευξη αυτού του αποτελέσματος. Η 9 Οκτωβρίου του 2017 η νέα προθεσμία και η ψηφοφορία στη Λίμπε θα γίνει στις 19. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά τα είπατε όλα. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια ακρόαση. Σας ευχαριστούμε και τους δύο για την εργασία σας ε, για αυτή την ε, οδηγία και το κανονισμό. Κύριε Μπόνι, θέλετε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Τερέζα. Με τη γνώση σου από την προηγούμενη θητεία σου στο Κοινοβούλιο και την εξέταση του θέματος και η αποφασιστικότητά σου τα τελευταία δύο χρόνια ήταν τους βασικούς παράγοντες. Και έτσι ολοκληρώνουμε το θέμα. Όλοι κατανοούμε, και είναι σημαντικό το αυτό, ότι περιέχονται πολλά σημαντικά στοιχεία για τα κράτη-μέλη, για τους Ευρωπαίους. Πρέπει να κατανοήσουμε όμως τις απειλές που αντιμετωπίζουμε λόγω των ναρκωτικών και των νέων ε, ψυχοτρόπων ουσιών. Όταν μιλάμε για ναρκωτικά, είναι πολύ επικίνδυνα, αλλά είναι ευκολότερο για τους γιατρούς να κατανοήσουν και να δώσουν κάποια θεραπεία όταν μιλάμε για τις νέες ψυχοτρόπες ουσίες, λόγω ελλείψεως ε, γνώσεων για τον αντίκτυπο στην υγεία μας, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, είναι δραματική κατάσταση. Δύσκολο να βρεθούν οι σωστές, οι ενδεδειγμένες θεραπείες. Χρειάζεται πολύ αυτή η οδηγία. Για να τεθεί τάξη στον τομέα. Και με τη συμμετοχή μας στο Κοινοβούλιο πρέπει να βρούμε τη σωστή προσέγγιση. Αυτό χρειαζόταν. Μας ενδιαφέρει το θέμα και είμαστε, αν θέλετε, και ε, το σημείο επαφής με τους πολίτες. Και τώρα και το, οι νέε λειτουργίε για το όλο το παρατηρητήριο είναι πάρα πολύ σωστά που αναφέρονται. Πρέπει να έχουμε ένα καλό σύστημα έγκαιρης προειδοποίηση. Χρειάζεται συνεργασία μόνο τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εντοπιστούν και να κατονομαστούν τα φαινόμενα και να υπάρχει και η βάση για την απαγόρευση κάποιων ουσιών σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Σκληρή μάχη δώσαμε με τα κράτη-μέλη. Μπορώ να το πω αυτό, πρέπει να το πω. Στο τέλος, λόγω των προσπαθειών της Μαλτέζικης Προεδρίας πετύχαμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ και πάλι Τερέζα, Πρόεδρος εργαστήκατε και ιδίω σκληρά. Και ευτυχώ αυτό αντικατοπτρίστηκε και στην ακρόαση την περασμένη εβδομάδα. Εργαστήκατε σιωπηλά, αλλά παρουσιάσατε τη σημασία του θέματος στο ακροατήριο την περασμένη εβδομάδα. Μας λείπουν κάποιοι σκιώδεις, δυστυχώς. Αυτό είναι το πρόβλημα με τις πέμπτες το πρωί. Αν δεν θέλει άλλο το λόγο, ευχαριστώ την Τερέζα για τη δουλειά που έκανα. 19 Οκτωβρίου η ψηφοφορία στη ΛΥΠΕ. Και ευχαριστούμε και τον κύριο Μπόνι. Και λόγω ημέρας και ώρας απουσιάζουν κάποιοι σκιώδεις. Συνάδελφοι, να πάμε στο επόμενο σημείο κατά αυτά είναι ο κύριος Βος. Πού είναι η πάλι του ΕΛΚ, γιατί δεν βλέπω φως. He's not answering his phone at the moment. We're working on it. I'm just relaying the messages.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 να αφήσουμε να πάρει ανάσα ο Άξελ, να ηρεμήσει, να χαλαρώσει. Ξέρω πολύ καλά ότι οι συνεδρίες της Επιτροπής πριν τις πληροφορίες της Πέμπτης δεν είναι η ιδεώδης διευθέτηση που δεν Ευχαριστώ όλα τα μέλη τα παρόντα, κυρίως αυτούς που ήρθαν από την αρχή. Και εργάζεστε σκληρά, Πέμπτη πρωί Στρασβούργο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βος που ήρθατε για 6 λεπτά νωρίτερα. Εσείς έρχεστε ακριβώς την ώρα σας, στο τσακ. Ευχαριστώ που ήρθατε νωρίτερα. Θα σας αφήσω να ανασάνετε, να κάνω μια εισαγωγή στο θέμα. Η υπηρεσία και η συνεργασία στα θέματα ποινική δικαιοσύνη των αρμόδιων φορέα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Εξέταση τροπολογιών για την πρόταση νέου κανονισμού για το Eurojust απόφαση του, την 187 του Συμβουλίου και που τροποποιήθηκε από την απόφαση 2009-46 και η πρόταση κανονισμού σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν για να αποκτήσει, να μπει στο πνεύμα της Λισαβόνας στο Eurojust και να αποκτήσει νέα διοικητική δομή. Ο κύριος Βος λοιπόν, αν είστε έτοιμος, παρουσιάστε το σχέδιο έκθεσης. μάλλον παρουσίασε το σχέδιο εκθέσεως τον Ιούλιο. Λάβαμε 232 τροπολογίες. Και τώρα θα αναφερθεί στις τροπολογίες. 12 Οκτωβρίου προβλέπεται η ψηφοφορία. Λοιπόν, Άξελ, μίλα μας στις τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ, Κλόντ. Και σας ευχαριστώ και όλους τους υπολείπους που με περιμένετε. Η πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον οργανισμό Eurojust είναι μια πρόταση του 2013 και έκτοτε τη συζητάει και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Στο Κοινοβούλιο ε, εμείς ε, λόγω και της νομοθετικής διαδικασίας έπρεπε να περιμένουμε τη συζήτηση του Συμβουλίου ε, και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γιατί γνωμοδοτούμε έτσι συνολικά για όλο το πακέτο. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και γι' αυτό. Όλοι οι σκιώδεις ακολούθησαν αυτή την πρόταση και την τακτική. Δεν ήθιστε, το ξέρω, αλλά μπορέσαμε, καταφέραμε να περιμένουμε έτσι ώστε να έχουμε μια συνολική έκθεση για να προσπαθήσουμε να την εγκρίνουμε συνολικά. Σας ευχαριστώ για την καλή συνεργασία και για την κατανόηση στα επιμέρους θέματα. Όπως είπες και εσύ, Πρόεδρο, στις 22 Ιουνίου ε, δημοσιεύτηκε η έκθεση τελικά. Συνολικά είχαμε 213 τροπολογίες που κατατέθηκαν και θα ήθελα να ευχαριστήσω και γι' αυτό, διότι ήταν πολύ επικοδομητικές οι ε, τροπολογίες αυτές. Άρα βρισκόμαστε στις συμβαστικές διαπραγματεύσεις και αύριο θα έχουμε μια δεύτερη τεχνική συνεδρίαση και η ψηφοφορία θα γίνει, όπως είπες και εσύ, στις 12 Οκτωβρίου. Έχει προγραμματιστεί. Τα πιο επίμαχα θέματα στον κανονισμό Eurojust είναι η προστασία των δεδομένων, αλλά και οι σχέσεις Eurojust με ε, την νεοσύστατη, που είπε και τη σύστασή της μάλλον την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για την προστασία των δεδομένων ε, σας είχα ε, πει ότι είχαμε τροπολογίες 97 τον αριθμό μαζί με τις δικές μου με πολύ διεστάμενες απόψεις. Εγώ ζητώ ε, να υπάρχει ρύθμιση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ξεχωριστή ε, ενώ για επιχειρησιακούς σκοπούς θα πρέπει αυτά να εξαιρούνται ενώ όλα τα άλλα στοιχεία και τα δεδομένα που αφορούν τη λειτουργικά ε, να ρυθμίζονται από την οδηγία 45-2001. Ε, οι άλλοι ζητούσαν όλα τα στοιχεία να περιλαμβάνονται σε αυτό το νέο σχέδιο του κανονισμού 45, κανονισμού 45-2001, όχι οδηγίες Αυτό ισχύει για όλους τους οργανισμούς, είναι ένας γενικός κανονισμός, ε, εισαγγελία Europol, Eurojust ε, όμως έχουν ε, μια πολύ ειδική ε, κατάσταση και χρειάζονται ειδικοί χειρισμοί και για τα προσωπικά δεδομένα και θα πρέπει να το βλέπουμε διαφορετικά από ό,τι για τους γενικότερους υπολείπους ε, οργανισμούς. Ε, έχουμε καταφέρει να καταλήξουμε σε μια συμβαστική πρόταση. Ε, έχουμε τακτές ανταλλαγές, ε, τακτικές ανταλλαγές απόψεων ε, και με την Κορνέλια Έρνστ που εκπονεί την έκθεση για την αναθεώρηση του κανονισμού 45 κάθετος 2001 που αφορά γενικά το χειρισμό των προσωπικών δεδομένων σε όλους τους οργανισμούς και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Για να καταλήξουμε όμως στο συμβιβασμό θα πρέπει αυτό που προτείνουμε να μην εμποδίζει την καθημερινή δουλειά και λειτουργία του Eurojust. Γιατί δεν το θεωρώ πρόοδο κάτι τέτοιο. Η ε, δικαστική και αστυνομική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντική για την αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος. Οπότε δεν θα πρέπει να τους δένουμε τα χέρια ε, και να τους βάζουμε τρικλοποδιές με τις υπερβολικές ρυθμίσεις. Τώρα, ποια είναι σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τα άρθρα 2, 3, 4 και 41 αναφέρονται και στην έκθεσή μου λέω ότι η ποινική δίωξη ε, θα πρέπει να συνεχίζει να γίνεται σε επίπεδο κρατών μελών ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Eurojust ε, θα πρέπει σεβόμενη την αρχή της αναλογικότητας και της επικουρικότητας να λειτουργεί. Ε, επίσης προσπάθησα να διευκρινίσω ότι μεταξύ Eurojust και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υπάρχει με ε, στενή συνεργασία, αλλά θα πρέπει να παραμείνουν και ε, ισότιμοι αυτοί οι οργανισμοί, αλλά και ε, ανεξάρτητη. Η Eurojust ε, λειτουργεί σε θελουσία βάση που τα κράτη-μέλη επιζητούν ε, την ε, συνεργασία της επαφές για τη διερεύνηση διασυνοριακών υποθέσεων. Ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να κινητοποιηθεί αυτεπάγγελτα στο πεδίο ορμοδιοτήτων της και αυτό είναι η συγκεκριμένη διαφορά. Άλλο Eurojust, άλλο Εισαγγελία θα πρέπει να ενισχυθούν και τα δύο και να συνδέουν έτσι ώστε όμως να μην υπάρχει σχέση προϊσταμένου-φυσταμένου. και η Eurojust να είναι ένα υποκατάστατο, μια βοηθητική υπηρεσία της εισαγγελία σε καμία περίπτωση. Έχουν ίδιες διακριτές αρμοδιότητες. Ε, τέλος όμως και αυτές οι συνδέσεις και οι σχέσεις της εισαγγελίας με Eurojust θα πρέπει να είναι σαφώς ορισμένες για να αποφύγουμε κενά, ελλείμματα ή επικαλύψεις. Το ίδιο ισχύει και για τη συνεργασία με τις χώρες εκείνες που δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ξέρετε ότι είναι 20 νομίζω τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, άρα μας λείπουν 8. Οπότε, τι θα γίνει με τους 8 αυτούς, άρα χρειάζεται πολύ σαφής ε, περιγραφή ε, του τι γίνεται και αρματιότητες. Έχουμε τροπολογίες ε, υπέρ της ενίσχυσης της Eurojust και κάποιες άλλες υπέρ της υποβάθμισης και της υπαγωγής στην εισαγγελία. Όχι. Είπαμε να είναι χωριστά, να υποστηρίζονται μεταξύ τους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν έχει σχεδιαστεί γι' αυτό το λόγο η εισαγγελία. Στις συμβαστικές κάνουμε κάποιες ε, προτάσεις πρόοδο και η Eurojust εδώ και χρόνια έχει αποδείξει ότι είναι αποτελεσματική και ε, υπάρχει και μεγάλη ζήτηση για τις υπηρεσίες της. Δεν θα πρέπει οι αρμοδιότητες της να περιοριστούν, αλλά να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα με την εισαγγελία. Να υπάρχει υποστηρικτική λειτουργία, αλλά διαφυλάσσοντας την ανεξαρτησία της Eurojust. Υπάρχουν και άλλες αρμοδιότητες, οι ποινικέ, έτσι κι αλλιώς είπαμε αυτά είναι των κρατών μελών, από εκεί εκπορεύονται. Μετά έχουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ασχολείται με την απάτη κατά των οικονομικών συμφερών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε και την εθελούσια δυνατότητα συμμετοχή στη Eurojust. Αυτά λοιπόν. Καταλαβαίνουμε ε, ε, ότι διαφυλάσσεται επικουρικότητα στα ποινικά θέματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Άξελ. Πολύ περιεχόμενο. Στου σκιώδει των σοσιαλιστών πάμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε έστω και αν ε, είναι κάπως ε, ατυχής η χρονική στιγμή αυτής της συζήτησης, πολιτικά ταιριάζει, γιατί ταυτόχρονα ε, ψηφίζουμε για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Άρα λοιπόν είναι καλό να συζητάμε σήμερα για την Eurojust. Αλλά λόγω του περιορισμένου χρόνου θα περιοριστώ σε λίγα σημεία. Το πρώτο ανέφερε ο κύριος Φως, ο κύριος Συγητής, αφορά την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Eurojust και εισαγγελία και νομίζω ότι αυτή είναι ένα θέμα, αυτό είναι ένα θέμα κεντρικής σημασίας και έχει την πλήρη μου υποστήριξη ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην υπάρξουν ούτε επικαλύψεις ούτε κενά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα ξεκινήσει τις εργασίες το 2020 και μέχρι τότε η Eurojust θα παραμείνει αρμόδια για την καταπολέμηση αξιόπινων πράξεων έναντι των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως πέρα από αυτό δηλαδή και πέρα από αυτά τα χρονικά όρια και σε εκείνες τις χώρες μέλη που δεν λαμβάνουν χώρα σε μια ενισχυμένη συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ένα δεύτερο σημείο που ανέφερε ο κ. Φως αφορά την προστασία των δεδομένων. Και εδώ θεωρώ ότι είναι πράγματι σημαντικό στο πλαίσιο τεχνικών συνομιλιών να θεωρώ ότι είναι σημαντικό το ότι πετύχαμε μια συμφωνία και ότι πράγματι το, όλη αυτή η θεματική ε, θα, θα πρέπει να ενταχθεί στο κανονισμό για την ε, ασφάλεια των δεδομένων, την προστασία των δεδομένων. Τώρα, ε, θα ήθελα να κάνω κάποιες κριτικές παρατηρήσεις. Πρώτον, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου το 2012 Υιοθετήσαμε μια κοινή θέση όσον αφορά τη δομή των ε, αποκεντρωμένων οργανισμών. Και και νομίζω ότι θα πρέπει να προσανατολθούμε σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να, η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπροσωπείται μαζί με δύο συναδέλφους και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο όργανο της Eurojust. Και θεωρώ ότι δεν, είναι, δεν θα πρέπει να εμπλακούμε πάρα πολύ στι λεπτομέρειε όσον αφορά τι δομέ τη Eurojust, γιατί γνωρίζουμε ότι η περισσία αυτή πραγματικά κάνει ένα πολύ καλό έργο και θα πρέπει να εμπιστευόμαστε τους εκπροσώπους της ότι μπορούν να ρυθμίσουν ορισμένα ζητήματα μόνοι τους και δεν χρειάζεται να συμπεριληφθεί μέχρι και τελευταία λεπτομέρεια στον κανονισμό. Τώρα, ένα ουσιαστικό πρόβλημα που αφορά την ψηφοφορία στις 12 του μηνός. Το είπε και ο Άξελ. Η δική μου εντύπωση είναι ότι δεν έχουμε προχωρήσει στις συζητήσει για τα κείμενα των συσβαστικών. Άρα θα πρέπει να περάσουμε και διαδράξουμε όλο το κείμενο. Σε ορισμένα δεν έχει γίνει καν κάποια διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να τηρήσουμε αυτή την υπερμηνία. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα, ότι ώστε να έχουμε ένα καλό κείμενο, να μην γίνει η ψηφορία στις 12 του μηνός για να έχουμε περισσότερο χρόνο να ασχοληθούμε με τις λεπτομέρειες. Δεν είναι άλλωστε και το, δεν και το τέλος του κόσμου. Ε, το θέμα αυτό ε, κρέμει εδώ και αρκετό καιρό και θα πρέπει να έχουμε την απαραίτητη ηρεμία να διευκρινίσουμε όλα τα ανοιχτά ζητήματα. Καλώς. Η Νάταλη είναι σκιώδης των φιλελευθέρων. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Κλοντ. Αγαπητοί συνάδελφοι, να πω κάποια πράγματα για την έκθεση. Σε έναν κόσμο όπου οι εγκληματίες αγνοούν τα σύνορα και οι, οι έρευνες για τα εγκλήματα πρέπει να προχωρούν όσο γρήγορα και εγκληματίες και να περνάνε τα εθνικά σύνορα. Αυτό το ζήτημα λοιπόν όσον αφορά την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του Eurojust έρχεται σε πολύ κατάλληλη στιγμή και ευχαριστώ τον Άξελ Βος για την έκθεση του που είναι πληρέστατη και για την πολύ σημαντική ακριβή μεθοδική δουλειά που έκανε στην προσπάθεια συγκερασμού των θέσεων στην παρούσα φάση επιδιώξεως συμβιβασμών όπως και η συνάδελφος Σιβών ε, ε, πρέπει να συζητήσουμε κάπως ίσως της, ε, την σύνταξη των συμβιβαστικών λαμβάνοντας υπόψη τις ευαισθησίες των ομάδες. Εν ονόματι της Άλτε εντάχει αναφερθώ σε τέσσερα στοιχεία που αντιστοιχούν στις τροπολογίες λίγο πολύ που καταθέσαμε. Πρώτον, χαιρετίζουμε το στόχο που είναι η αποσαφήνιση που έγινε μέσω εργασία των νομικών, το τόνισε ο Άξελ Βός, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για να καθοριστούν σαφέστατα οι αρμοδιότητε, η περίμετρος αν θέλετε, του κάθε στοιχείου που περιέχεται για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Η ομάδα μου, όπως έδειξε από τις κατευθύνσεις τροπολογίε, επιμένει να διευκρινιστεί πολύ καλά η σχέση μεταξύ Eurojust και της Ευρωπαϊκής Αγγελίας η διάρθρωση μεταξύ των δύο φορέων, όπως αναφέρθηκε από τους συναδέλφους. Και όταν θα εμπλέκονται τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στον κύριο Τζόστ, αλλά όχι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και ελπίζουμε να, να συμμετάσχουν αυτοί που δεν συμμετέχουν. Και όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Κάτι άλλο που δεν θα εκλούσει συναδέλφους. Η ομάδα μου επιθυμεί διακαώς αυτός ο οργανισμός να έχει το μεγαλύτερο δυνατό ευρωπαϊκό χαρακτήρα, κοινοτικό χαρακτήρα του ΣΥΠΗΝ. Του δίνουμε μεγάλη σημασία. Και η δυνατότητα πρωτοβουλίας που προβλέπει τις συνθήκες πρέπει να ενισχυθεί. Η πρότασή μας δεν τη χάνει στη ρήξη της πλειοψηφίας. Χρειάζεται επεξεργασία το θέμα. Γιατί το λέμε αυτό από τις συζητήσεις τι διαπιστώνουμε και τις εργασίες μας. Μεταρρυθμίζουμε τρία-τέσσερα χρόνια μετά ένα νομοθέτημα που χρειάστηκε τέσσερα χρόνια για να επικαιροποιηθεί και γίνεται απερχαιωμένο πάρα πολύ γρήγορα. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερα ευρωπαϊκά μέσα και εργαλεία για να αποφύγουμε αυτού του είδους τα προβλήματα πρέπει να ακολουθήσουμε κοινοτική προσέγγιση στο βαθμό του δυνατού. Και κάτι πολύ σημαντικό για την ομάδα μου, αυτό που θα αναφέρω. Το εφαρμοστείο καθεστώ για τα προσωπικά δεδομένα από πλευρά Eurojust, πώ θα τα επεξεργάζεται. Στο 40, κανονισμό 45-2001 προβλέπεται κάτι τέτοιο. Αναθεωρείται βέβαια η σχετική διάταξη. Καθορίζεται ένα ενίο καθεστώ προστασία προσωπικών δεδομένων για όλα τα θεσμικά όργανα. Θα ήταν καλό να εφαρμοστεί αυτό να μην έχουμε εμβαλωματικέ λύσει όπου κάθε φορέα, κάθε οργανισμό διέπεται από διαφορετικό καθεστώ και έχουμε πολυμορφία καθεστώτων. Και ωραία δεν είναι και περίπλοκη είναι και δεν θα είναι και αποτελεσματική μια τέτοια λύση. Τέλο, τέταρτο σημείο. Ε, δείχνουμε μεγάλη ευαισθησία να αφορά τον επιδιωκόμενο στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Δηλαδή, να υπάρχει ταχύτερη δικαστική συνεργασία στην Ευρώπη να βελτιωθεί άρα και η αποτελεσματικότητα του οργανισμού. Να πούμε δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Καταθέσαμε τροπολογίες σχετικές. Υποστηρίζουμε τη διευκρίνηση της δομής του Eurojust. Διάκριση μεταξύ του Ομοδίου Σώματος για επιχειρησιακά θέματα και του Εκτελεστικού Συμβουλίου για όλα τα θέματα, τα διαχειριστικά και διοικητικά. Αυτά είναι τέσσερα σημεία, επ' αυτόν επιμένουμε. Και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον Άξελ Βος. Έξοχη η συνεργασία μας και θα συνεχιστούν οι συζητήσεις επί του θέματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Νάταλη. Τέλος. Εύα Ζολή και μετά ο συγγητής. Ζολή. Ευχαριστώ Κλοντ που μου δίνεις το λόγο. Ευχαριστώ και τον Άξελ Φως για την εξαιρετική του εργασία σε αυτό το θέμα. Συμφωνώ με τους υπολείπους και όδες ηγητές. Ε, να πω ότι και η δική μου πολιτική ομάδα ενδιαφέρεται πάρα πολύ ε, γρήγορα να στηθεί ε, αυτός ο οργανισμός. Αλλά 12 του μηνός είναι μάλλον πολύ γρήγορα για να ψηφίσουμε γιατί είναι σημαντικό θεσμικό όργανο και χρειαζόμαστε ακόμα κάποιες προσαρμογές να κάνουμε για τη διαρθρωτική συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τον οργανισμό Eurojust. Η δική μου λοιπόν πολιτική ομάδα τη φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να ενημερώνεται και να ενέχεται πλήρως στις υποθέσεις Eurojust που μπορεί να την αφορούν. Αυτό ε, εκφράζεται με δικαίωμα ψήφου της εισαγγελία ε, στο κολέγιο του Eurojust, ε, όταν πρόκειται πάντα για θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η συνεργασία των δύο θεσμών αυτών θα πρέπει να είναι ειλικρινής και ουσιαστική. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι ε, μπορούμε να πιστευτούμε την καλή πίστη και τη βούληση των κρατών μελών για την εθελοντική του συμμετοχή, τουλάχιστον στην αρχή. Ε, άρα είναι πολύ σημαντικό να καταστήσουμε υποχρεωτική ε, την ενημέρωση της ε, εισαγγελίας από πλευράς Eurojust. Δηλαδή να είναι δεσμευτικό και όχι να εναπόκειται στον πατριωτισμό των κρατών μελών. Επίσης, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το καθεστώς προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Υπάρχουν ε, ήδη ε, διάφορα ε, καθεστώτα που είναι ενιαία και αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν και όχι να εφεύρουμε κάτι ειδικό και ιδιαίτερο για τη Eurojust. Νομίζω ότι είναι ευρία η συμφωνία και υποστηρίζω αυτά που είπαν οι υπόλοιποι σκιώδεις, ιδιαίτερα η Ναταλή Γκρισμπέκ. Ευχαριστώ. Λάουρα, γρήγορα, παρακαλώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή, τον Άξελ Βος, έξοχη δουλειά που έκανα Με τις τροπολογίες θα εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου στη διακυβέρνηση του οργανισμού. Σύμφωνα με πρόσφατες διατάξεις που θετήθηκαν για άλλους οργανισμούς ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και οι σχετικέ ρυθμίσει τροποποιήθηκαν πρόσφατα. Έχουμε κοινή δήλωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ε, του 2012 για του οργανισμού. Ζητούμε ο Πρόεδρο να επιλέγεται από υποψηφίου που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά διαδικασία επιλογή που θα είναι ανεξάρτητη και θα βασίζεται επί δεξιοτήτων και γνώσεων και θα πρέπει να εμφανίζονται στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών οι υποψήφοι και θα γνωμοδοτεί και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη όσον αφορά τον διορισμό του Προέδρου αυτή τη γνωμοδότηση. Ήταν θέλουμε συνεργασία αποτελεσματική μεταξύ Ευρωπαϊκή Αγγελία και Eurojust, λαμβάνοντα υπόψη τι ιδιαιτερότητα τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Κάτι που θα ψηφίσουμε σήμερα. Και όσον αφορά την προστασία των δεδομένων που θα εφαρμόζεται για τον οργανισμό, θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τον κανονισμό το γενικό σαν την προστασία των δεδομένων και πιο συγκεκριμένα το καθεστώ θα πρέπει να είναι αυτό που προβλέπεται από τον κανονισμό 45 του 2001. Και από αυτό ευχαριστώ τον εισηγητή για την ευελιξία που επέδειξε, αποδεχόμενος να παραπομπεί τον κανονισμό 45-2001 και ελπίζω οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται την αναθεώρηση του κανονισμού να ολοκληρωθούν σύντομα. Εν γέννη, Πολλά έγιναν για να πετύχουμε μια συμβαστική λύση αποδεκτή από εμά, όμως απομένουν κάποια σημεία προς διευκρίνηση. Είμαστε διαθέσιμοι να ακολουθήσουμε την προσέγγιση του συγκητή που έχει σαν στόχο να υπάρξει σαφής διάκριση όσον αφορά τη δομή της διακυβέρνησης του οργανισμού μεταξύ επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων και πραγματικά διοικητικών αρμοδιοτήτων ε, η ε, υπερβολική απλούστευση όμως θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη, θα μπορούσε να δημιουργήσει αβεβαιότητα όσον αφορά τη διαχείριση του οργανισμού. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε, να καθορίσουμε ποιε πρέπει είναι οι αρμοδιότητε για τι οποίε είναι υπεύθυνο ε, ο οργανισμό. Είμαστε διαθέσιμοι για να καταλήξουμε σε κάποιο συμβιβασμό και εύχομαι καλή δουλειά στον ε, εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ, Λάουρα. Ευχαριστώ. Θα πιστέψω στον εισηγητή και ευχαριστώ τα μέλη για την ποιοτική, πολύ ποιοτική συμμετοχή στις προσπάθειες του εισηγητού. Δεν τα καταφέρνουν αυτό ε, λίγα λεπτά από τις συμφορίες ε, της Πέμπτης στο Στρασβούργο ή άλλες επιτροπές. Ευχαριστώ που παρίσταστε εδώ. Τα καταφέρνουμε σαν Λίμπε και πρέπει να γίνονται η συνεδριάσει για να τηρούμε το χρονοδιάγραμμα. Και συγγνώμη που συνεδριάζουμε πριν τι ψηφοφορίε. Άξελ, δεν θα έχουμε χρόνο να απαντήσει όλα τα σημεία ενδελεχώ. Ίσως να αναφέρεις την άποψή σου για την ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα. Αν μπορεί ε, να τοποθετηθεί επ' αυτού θα βοηθούσε. Καταρχά, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους και όπως και ο Πρόεδρος για τις συνομιλίες και τις ανταλλαγές που είχαμε συμφωνώ απολύτως για τα επιμέρους θέματα ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αναβολή της ψηφοφορίας δεν έχω πρόβλημα εγώ καταρχήν και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην ποιότητα και όχι στην ταχύτητα αλλά ε, να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να προχωρήσει όσο για αυτό το πράγμα να βολιδοσκοπήσουμε τι δυνατότητες έχουμε χρονικές, ε, τι προτείνει η Προεδρία, γιατί ήθελε να προχωρήσει, ε, να δούμε πώς έχουν ε, οι δυνατότητες, αν υπάρχει ευελιξία. Παρακαλώ τον Πρόεδρο να το κοιτάξει. θα σας τα θα συνεννοηθούμε με τους σκιώδης ηγητές τι δυνατοτητε εχουμε έχουμε. Δύο-τρία πράγματα. Είναι σημαντική η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Βεβαίως, πάντα έχουμε την επιλογή να πούμε κάνουμε κάτι διαφορετικό για τη Eurojust ή ε, κινούμαστε στην άλλη οδηγία κανονισμό, τι είναι, δεν θυμάμαι, 45 το 2001. Ε, αλλά έχουμε και τα θέματα για την αστυνομία και τη δικαιοσύνη ε, για την προστασία δεδομένων όταν τα χειρίζονται ιδιοκτικές αρχές. Η δική μου πρόταση ήταν να ε, προσαρμοστούμε στη Europol και ε, να το μεταφέρουμε περίπου στη Eurojust. Αυτή ήταν η πρόθεσή μου. Είμαι στη διάθεσή σας όμως. Αν έχετε μια άλλη πρόταση να το δούμε, λογικά να καταλήξουμε κάπου και να τα συμπεριλάβουμε αυτά τα θέματα. Δύο-τρία ε, πράγματα μόνο για το δικαίωμα πρωτοβουλίας και ε, της Eurojust. Έτσι αλλοιώνουμε ε, την ίδια τη χρειά και τη φύση αυτού του οργάνου γιατί αυτή τη στιγμή λειτουργεί εθελοντικά. Δηλαδή τα κράτη-μέλη έρχονται και απευθύνονται στη Eurojust και ζητούν διασυνοριακές διώξεις, έρευνες κτλ. Τώρα, αν έχει δικαίωμα ίδιας πρωτοβουλίας, δηλαδή αυτεπάγγελτα να δρά ψυχολογικά αυτό στα κράτη-μέλη οδηγεί σε αγγυλώσεις. Ε, να τρέχουν λιγότερο ε, στη Eurojust για να εκμεταλλεύονται τη συνεργασία ε, γιατί ψυχολογικά θα φοβούνται ότι θα τους πάρουν την αρμοδιότητα και θα χάσουν τον έλεγχο. Λίγη επιφύλαξη και συγκράτηση συνιστώ. Αυτή είναι η φύση η ίδια της Eurojust αυτό το εθελοντικό το δέχονται τα κράτη-μέλη και αυξάνονται και οι αριθμοί και το δείχνουν να μην τους αναγκάσουμε να μην τους το επιβάλλουμε. Και είναι γενικά διάφορες δομές, όχι μόνο στο εσωτερικό της Eurojust, είναι το κολέγιο και το εκτελεστικό ε, συμβούλιο ε, υπάρχουν μετά τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που δεν συμμετέχουν, η Europol και η ίδια εισαγγελία. Τι σχέσει έχουν μεταξύ τους όλα αυτά σε συγκεκριμένο στερέωμα. Αν καταφέρουμε να τα ρυθμίσουμε νομίζω θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Για το χρονοδιάγραμμα, πρόεδρο, βεβαίω. Ε, ρίχνει τον παλάκι στον Πρόεδρο. Παρακαλώ, από ό,τι φαίνεται ε, ήθιστε, ε, δεν πειράζει, να το φροντίσω. Αύριο υπάρχει μια τεχνική συνεδρία σε επίπεδο υπαλλήλων, να δούμε τι δυνατότητες έχουμε. Ε, γιατί είναι και πολύ σφιχτή ημερήσια διάταξη για την άλλη εβδομάδα. Να δούμε αύριο τι επιλογές υπάρχουν. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να διατηρήσουμε την ποιότητα του θέματος αυτού. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, ε, είναι πολύ σημαντικό. Εχθές είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ολομέλεια. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει αύριο στη συνεδρία σε αυτή των υπηρεσιακών παραγόντων και θα προχωρήσουμε. Και εγώ το ε, αναλαμβάνω να κοιτάξω για την απόφαση που θα πάρει. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και για την πειθαρχία που δείξατε σήμερα το πρωί. Λήξη συνεδρίασης, επόμενη συνεδρίαση 11 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε.